Also Ας ξεκινήσουμε και πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη, θέλω να χαιρετήσω μια ομάδα από τον Γκαμπριέ, επισκεπτών από την... που έχει φέρει ο Γκαμπριέλ Κρόνης. Έρχεστε από την δική μου ιδιαίτερη εκλογική περιφέρεια και θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω ιδιαίτερα εδώ στις Βρυξέλλες από την περιοχή της Βόρειας Ινανίας Βεσφαλίας. Και τώρα για την ημερήσια διάταξη χαιρετίζω την παρουσία του συναδελφού μας του κυρίου Γιέντς Γκάιερ που είναι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Έχουμε παραδοσιακά πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο κύριος Γκάιερ θα αναφερθεί στις προτεραιότητες και στην κατάσταση του προϋπολογισμού του 2017 και θα έχουμε μετά ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Είναι σημαντικό οι προτεραιότητε τη. Ε, Επιτροπής μας να αντανακλώνται και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ώστε το Κοινοβούλιο έναντι του Συμβουλίου να μπορεί να έχει μια στεναρή στάση για τον προϋπολογισμό του 2017. Σας δίνω λοιπόν κύριε Γκάιερ τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Μιχαήλ, εγώ είμαι από την <laughs> ΕΣΥ βεβαίως. Σα Σας καλωσορίζω κι εγώ. Γείτονες είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι τα λεφτά λοιπόν. Οπότε φαντάζεστε πως όταν μιλάμε για το πώς θα ξοδευτούν, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις και πώς θα ε, έχουν τα πράγματα, ίσως να είναι η συμμετοχή λιγότερο να είναι κάπως μικρότερη από ό,τι στις ε, ψηφοφορίες για το πώς θα ξοδευτούν. Λοιπόν, ήμουνα στην Επιτροπή Ισότητας ε, σήμερα το πρωί και θεωρώ πως ε, όλοι θα μου πούνε ότι ναι πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες ε, αλλά εμείς είμαστε πιο σημαντικοί. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα δυσαρεστήσω πολλούς. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίναμε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμμετείχαν οι συνάδελφοι. Αυτές είναι οι προτεραιότητες θα έλεγα και η γενικότερη εκτίμηση των προβλημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς έχει ο προϋπολογισμός 2017 και είμαστε σε μια πολύ επισφαλή θέση. Όλοι πολιτικοί είμαστε εδώ μέσα, οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαφορετικές κρίσεις. Δεν θα τα ξαναπώ. Οπότε η κατάσταση αυτή μας οδηγεί στο ότι στις προηγούμενες διαβουλεύσεις ε, για τον προϋπολογισμό 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που υπάρχουν στον προπολογισμό με μία εξαίρεση το λεγόμενο περιθώριο ανάγκης στο οποίο αν βάλουμε χέρι θα πρέπει να επιστρέψουμε τα λεφτά μέχρι το 2020. Οπότε, αν ε, τα ξοδέψουμε θα πρέπει να τα βρούμε κάπου αλλού τα επόμενα χρόνια. Όλα τα άλλα μέσα τα χρησιμοποιήσαμε και η κατάσταση της κρίσης δεν άλλαξε. Αντιθέτως επιδεινώθηκε. Χτες στο νεαρινό τριμερή διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα συμφωνήσαμε ήδη τον πρώτο τροποποιητικό προϋπολογισμό η κινητοποίηση 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε ένα νέο πολιτικό μέσο για το οποίο συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, αλλά βεβαίως το θέμα είναι πόσο θέλει το Συμβούλιο, για πόσο καιρό θα συνεχίσει να παίρνει λεφτά από τον περιπολογισμό για να μπορεί να λύνει όλες αυτές τις νέες καταστάσεις που οπωσδήποτε είναι επίουσες. Δηλαδή 270, κατάσταση, 270 εκατομμύρια πλέον για την κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία που πρέπει να βρεθούν το 2017 και μάλιστα από τον προϋπολογισμό που αποφασίσαμε και έχουμε επιπρόσθετες δαπάνες. Αν υποθέσουμε πως η ανθρωπιστική κατάσταση θα εξακολουθήσει να είναι δύσκολη, θα χρειαστούν και άλλα κονδύλια. Για να μην σκεφτούμε ότι θα γίνει να προκύψει καμία άλλη κρίση στη Γεωργία ας πούμε. Έχοντας αυτά κατά νου. Καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, το Ευρωπαϊκό αυτό κοινοβούλιο θέλει να χρησιμοποιήσει τον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να κάνει πολιτική για τους ανθρώπους, για την κατάσταση την κοινωνική, του περιβάλλοντος και τα αλλά πρέπει να είναι σαφές πως ε, τα ε, κονδύλια μας είναι πολύ περιορισμένα. Και Βεβαίω, γνωρίζουμε πως αυτά τα πράγματα δεν είναι δωρεάν και είχατε εκφράσει την αντίρρησή σας για το ότι αφαιρέθηκαν χρήματα ακριβώ ειδικά από το Connecting Europe Facility με το οποίο θέλετε να κάνετε συγκοινωνιακή πολιτική. Και αντιλαμβάνομαι την δυσαρέσκειά σας, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου το εξή. Το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει το ποια θα είναι τα λεφτά Στη νύχτα αυτή των μεγάλων μαχαιριών, όπως ε, την λέω, όταν μαζεύτηκαν 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και συμφώνησαν στο δημοσιονομικό πλαίσιο, η κάθε χώρα πήρε τον λεγόμενο εθνικό φάκελο που περιγράφει αφενός ε, πόσα λεφτά πληρώνει, συνεισφέρει στον προπολογισμό η κάθε χώρα, αλλά περιγράφει και αντιστρόφως πόσα λαμβάνει από τα κοινωνικά ταμεία, περιφερειακά ταμεία, τα γεωργικά ταμεία και τα λοιπά ταμεία. Και τα κράτη-μέλη έβγαλαν το συμπέρασμα από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και είπαν πως θα ε, εξετάσουν στη μέση του διαστήματος αυτού εάν παραμένουν άθικτοι αυτοί οι εθνικοί φάκελοι. Το κοινοβούλιο διαφώνησε, αλλά ήταν κάτι το οποίο είχαμε χάσει στη συνθήκη της Λισαβόνας, ένα από τα λίγα μειονεκτήματα που είχαμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν όμως γίνει αυτό, σημαίνει πως η Κομισιόν θα έχει πολύ λιγότερα λεφτά για να τα διαθέσει όπως θέλει και για να χρηματοδοτήσει το ΕΦΣΕ. Οπότε αφενός θα περικοπεί η χρηματοδότηση της έρευνας και το Connecting Euro Facility γιατί δεν έχει και εθνική συγχρηματοδότηση και δεν πρέπει να έχει. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα και μετά έχουμε την δεύτερη άσχημη είδηση. Από τα 8 δισεκατομμύρια πρέπει να κινητοποιήσουμε, έχουμε μόλις τα 3,3 και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινητοποιηθεί για να βρει τα υπόλοιπα. Και φοβάμαι πως η Κομισιόν δεν θα έχει καμιά καλύτερη ιδέα φέτος. Εμείς ως Επιτροπή του Προϋπολογισμού θα κάνουμε ό,τι κάναμε και πέρσι. Δηλαδή, θα ακολουθήσουμε την ε, ψηφοφορία της ε, Επιτροπής σας ε, έτσι ώστε όταν απαιτηθεί να ξαναφύγουν λεφτά από το ΕΦΣΙ και των Ταμείων των Μεταφορών να το επισημάνουμε αναλόγως ε, στη δική μας την ψηφοφορία. Βεβαίως δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα, με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν τα κονδύλια. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Και να σας πω πως και η Κομισιόν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, οπότε η διαπραγματευτική μας θέση, δηλαδή δεν μπορούμε να προτείνουμε και κάπου εναλλακτικά από όπου μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Αν έχει κάποιος κάποια ιδέα, σας παρακαλώ. Και θα είμαι ευγνώμων. Δεν μπορώ λοιπόν σήμερα να σας υποσχεθώ ότι θα έρθω μετά τη διαπραγματεύση να σας πω ότι τα καταφέραμε. Ορίσαμε λοιπόν προτεραιότητες οι οποίες βεβαίως σχετίζονται όχι μόνο με τις επίκαιρες κρίσεις αλλά και οι άλλες κρίσεις που είχαν προβλέψει δεν έχουν επιληθεί. Δεν υπάρχει επαρκής καινοτομία. Υπάρχει ακόμα πολύ υψηλή ανεργία, υψηλή ανεργία των νέων και επιπλέον έχουμε τους στόχους ε, της ε, Ευρώπης 2020 Όλα αυτά είναι στις ε, κατευθυντήριες γραμμές του προπολογισμού. Και, ξαναλέω, ειδικά στην καταπολέμηση της φτώχειας είχαμε πει ότι η παιδική φτώχεια είναι μια ιδιαίτερη μορφή που πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, ότι είναι ένα φαινόμενο δηλαδή που πρέπει να μας αναγκάσει να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο φτώχειας των πιο ευπαθών της κοινωνίας μας. Έχουμε λοιπόν πλευρή κρίση, χωρίς να έχουμε περισσότερα κονδύλια. Οι ανάγκες χρηματοδότησης αυξάνονται και τα κράτη-μέλη δεν έχουν καμία όρεξη να δώσουν περισσότερα λεφτά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Οπότε συνεχώς στις διαπραγματεύσεις μας λένε ότι πρέπει να υπάρξει μια σύνθεση με την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου μουσιονομικού πλαισίου και οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πιέσει για να χρησιμοποιηθεί αυτό. Δηλαδή να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με αυτά και θα πούμε ότι όχι, αν είναι να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, που μας έχουν αναθέσει τα κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ. Τώρα τον λόγο έχει η Ιζαμπέλα Ντεμόντη, η συγγητριά μας. Ε, Ευχαριστώ. Με ευχαριστήσω που συγγείτε καταρχήν για τι κατευθυντήρες γραμμέ που μα έδωσε για τον προπολογισμό του 2017 και να υπογραμμίσω κάποιε πτυχέ. Καταρχά, πολύ σωστά υπόθηκε ότι υπάρχει μια συρρήκνωση σε μια κατάσταση κρίση. Ακριβώ γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσει που θα δημιουργούσουν θέσει απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, θα διευκολύνουν το εμπόριο, τις μικρομεσαίε επιχειρήσει και τι επενδύσει ε, διασυνοριακά. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί στο άρθρο 10 έβαλε και το CEF, το Connecting Europe Facility, που είναι ένας μηχανισμός απαραίτητος και πολύ σημαντικός που θα αντισταθμίσει τις περικοπές. Όπως υπόθηκε πριν από λίγο, αυτές οι περικοπές είναι πολύ ουσιαστικές. Και αυτό που είχαμε πει και στο παρελθόν ήταν να υπάρχει κάποιο αντιστάθμισμα, ούτως ώστε να υπάρξει μια μόχλευση των... Μάλλον, ε, το φαινόμενο της μόχλευσης για αυτά τα ταμεία, για τα κονδύλια από αυτά τα ταμεία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε χώρο και στον τουρισμό που είναι τομέα κλειδί για την οικονομία. Έχει δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και βοηθάει για να, καταπολε... να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων κυρίως, που είναι σε δραματικά επίπεδα. Την ανεργία των νέων και των γυναικών. Και να δώσει κάποιο περιθώριο σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία. Τις απομακρυσμένες περιοχές ας πούμε και μπορεί να δημιουργήσει κάποια ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί. Ε, σε όλους τους τομείς των μεταφορών δεν θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές στις χρηματοδοτήσεις για μέτρα υπέρ της ασφάλειας. Θα πρέπει από την άλλη όμως να υπάρχει και μια δημοσιονομική διαφάνεια για όλες τις ε, υπηρεσίες, για όλους τους οργανισμούς. Τώρα για τον τουρισμό, να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε, ε, να χρησιμοποιήσουμε πολύ ε, τα μια τα επενδυτικά, να έχουμε δηλαδή υψηλή χρηματοδότηση από αυτά και να υπάρξουν και πιλωτικά προγράμματα, πιλωτικά σχέδια τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία. Γιατί αυτή είναι η προπαρασκευαστική φάση και είναι σημαντικό για να φτάσουμε σε πραγματικά προγράμματα επενδύσεων ε, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από διαγωνισμούς κτλ. Ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις σκέψεις του εισηγητή. Είχα και την ευκαιρία μάλιστα να συνεργαστώ με τον κύριο Γκάιερ για μία έκθεση με την οποία ε, ασχολήθηκα εγώ και εκείνος τότε ήταν ε, σκιώδης εισηγητής. Και με αυτή τη συνεργασία είδαμε ότι μπορεί ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι ε, που θα συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Τα δικά του, τα δικά μου δηλαδή. Σε αυτήν την περίπτωση μιλούσαμε για τους εταιρικού φόρους. Τώρα, ε, κάτι που είπε ο συγητής και η προλαλήσασα. Καταρχάς, με θλίψη διαπιστώνω ότι οι ελλείψεις πόρων για το ΕΦΣΥ θα αναγκάσουν την Κομισιόν να προτείνει ε, επιπλέον περικοπές ε, στο ΣΥΕΦ. Αυτό με αναγκάνει, αναγκάζει να εξάσω την εξή ε, σκέψη που ελπίζω να γίνει αποφασιστικό για την ε, πρόταση του προπολογισμού. Δηλαδή, να αξιολογήσουμε πραγματικά τις επιδόσεις των ε, μέσων που έχουμε στην διάθεσή μας. Γιατί το CF, όπως είναι γνωστό, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται κανονικά για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις στον τομέα των υποδομών των, των μεταφορών. Αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί καλά πάνω απ' όλα ε, μοιάζει τετριμένο, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά παρεμβαίνει εκεί ακριβώς όπου είναι δύσκολο να βρούμε πόρους, ιδιωτικούς πόρους, για να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Και αυτό είναι το περίεργο όλη αυτής της ιστορίας ε, με τη μεταφορά πόρων από το CF στο ΕΦΣΙ. Όπως είπε και, η Δεμόντι, έχουμε δύσκολη μόχλευση στο ΕΦΣΙ και αφαιρούμε πόρους από το CF το οποίο χρηματοδοτεί ακριβώς αυτές τις επενδύσεις που δεν, έχουν, ε, δεν υπάρχει εύκολη μόχλευση και δεν κινητοποιούνται εύκολα τα ιδιωτικά ε, κονδύλια, τα ιδιωτικά κεφάλαια. Φυσικά όλα αυτά που είπατε, που καταγγέλλετε, είναι σωστά. Από την άλλη όμως αυτή η μεθοδολογία, ας πούμε, μεταφοράς πόρων από το ΕΦΣΙ στο CF, είναι μεθοδολογικά λάθος. Δεύτερον, τουρισμός. Πρέπει να μιλήσουμε για τους πόρους. Η Ιζαμπέλα Ντεμόντε μίλησε για το κόσμο και εγώ θέλω να προσθέσω ένα στοιχείο που έχει έτσι πολιτιστικό χαρακτήρα και ως Ιταλός θα το πω έτσι. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον τουρισμό ως εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης. Σκέφτομαι την Ιταλία τώρα, έτσι. Εμείς κάποτε δεν ήμασταν... Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποτε είμαστε φάνταστοι, δημιουργικοί και τα λοιπά και τώρα πάψαμε να είμαστε. Όχι, είμαστε ακόμα. Ερχόμαστε, έρχονται διάφοροι Ασιάτες, ε, ε, Κινέζοι και τα λοιπά έρχονται σε εμά για να δουν πώς φτιάχνουμε ας πούμε διάφορα πράγματα στην βιομηχανία και γυρνάνε πίσω και τα εφαρμόζουν αυτά που βλέπουν. Αυτά ήθελα να πω χοντρικά για έτσι, αδρές γραμμές για αυτό το προπολογισμό. Παύελ Τελέσκα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ, τον εισηγητή. να ξεκινήσω με μια γενικού χαρακτήρα παρατήρηση. Δεν μου είναι ευχάριστο που το λέω αυτό. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω ότι μπορούμε να καφηθούμε για πολλές επιτυχίες. Ιδίως και στον τομέα μας. Αν δούμε τα τελευταία 5, 7, 8 χρόνια, αν υπάρχει κάποια επιτυχία, που υπήρχε στην πολιτική μας ήταν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT. Έχουν αποδώσει καρπούς που είχαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Μια δεύτερη παρατήρηση. Ίσως είναι πολύ αργά να κλαίμε πάνω από το χειμένο γάλα, αλλά η Κομισιόν με την πολιτική μας <clears throat> υποστήριξη επινόησε το εύση. Τι είναι το εύση όμως είναι μια πρωτοβουλία ώστε να δημιουργήσει ιδιωτικέ επενδύσεις και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει την απασχόληση, να δημιουργήσει απασχόλησης. Αλλά σε βάρος του, των TNT και άλλων σχεδίων που είναι επίσης δημόσιας χρηματοδότησης υπάρχουν ε, έργα όπως η Ρία Μπάλτικα που μόνο χάρη στην χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό ισχύει και για πολλά άλλα σχέδια και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν είναι μονάχα να διατηρήσουμε τους πόρους στο ΕΦΣΥ για τις μεταφορές, αλλά να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετική η φύση των σχεδίων και διαφορετική η δικαιούχη, στο ΕΦΣΥ και ο ηγητή καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι το, για το οποίο μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά επειδή θέσατε την έμφαση <clears throat> για αυτά τα σημεία, θέλω και εγώ να το υπογραμμίσω. Επομένω, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, δηλαδή πρέπει να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τη χρηματοδότηση του ΣΕΦ, του Connecting Europe Facilities, και για ένα άλλο λόγο, γιατί πολλά από αυτά τα σχέδια είναι ήδη εν εξελίξη. <clears throat> Αν σταματήσουμε τη χρηματοδότηση θα αυξήσουμε το συνολικό κόστος της χρηματοδότησης. Αν κόψουμε ή αν καθυστερήσουμε αυτά τα σχέδια, τότε <clears throat> θα κοστίσουν συνολικά πολύ περισσότερο. Και αυτό δεν έχει να κάνει μονάχα με τον οικονομικό κύκλο, αλλά φυσικά και αυτός ο οικονομικός κύκλος παίζει κάποιο ρόλο. Θα συνεργαστώ λοιπόν εγώ με μεγάλη χαρά με τον συγητή και με τους κοιόδης εισηγητές για το θέμα αυτό και δέχομαι την ε, πρότασή σας, την πρόκλησή σας να έρθουμε με ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε δημιουργικοί για να κάνουμε πιο εύκολη τη δική σας ζωή, αλλά και να πετύχουμε να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες μας. Πράγματι λοιπόν θα προσπαθήσω να επανέλθω με προτάσεις. Τώρα βέβαια, εγώ δεν είμαι Ιταλός, αλλά μας ενδιαφέρουν και τα θέματα των μεταφορών και του τουρισμού. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση στο γεγονός ότι και ο τουρισμός είναι πηγή ε, πλούτου και ανάπτυξης. Επίσης αναφερθήκατε κύριε Ισηγητά σε πολλές κρίσεις και προσυπογράφω όλα αυτά που λέτε. Και υπάρχουν και άλλες κρίσεις που θα μπορούσε κανείς να αναφέρει. Ας ε, κρατήσουμε όμως κάποια αυτοπιθαρχία, όχι εσείς, όχι εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών. Αλλά να σκεφτούμε για τα κρατημέλη που έχουν έργα στη δική τους αρμοδιότητα καταρχήν, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν βολευτεί με τη λογική ότι πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρηματοδοτεί. Εμείς θέλουμε να έχουμε κοινέ πολιτικές, μια από τις οποίες είναι η πολιτική μεταφορών. Όλα αυτά λοιπόν που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης και είναι κοινέ πολιτικές και διαμεθοριακού χαρακτήρα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και να είναι πιο επιλέξιμα στα, για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι οι κρίσεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη μας έχουν συνηθίσει σε αυτή την πρακτική θέματα δικής του αρμοδιότητα τελικά να καλύπτονται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αυτά τα ίδια θα έπρεπε να κάνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και μπορώ να επανέλθω σε πιο πολλές λεπτομέρειε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Δεκιο Πρώτο. Η Καρίνα Ντέλη. Ευχαριστώ. Άκουσα τον εισηγητή με προσοχή Αλλά δεν μας δώσατε έτσι και ένα φιλοπορίας, δηλαδή τις διάφορες πάσεις, ημερομηνίες για τα πιλωτικά σχέδια, για τις προπασκευαστικές δράσεις κτλ. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να μας δώσετε όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές τις πληροφορίες. ich habe mich jetzt auch zu Wort gemeldet. Λοιπόν, και εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Αναφερθήκαμε σε τρεις ε, στόχους. Αντιμετώπιση της ανεργίας, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κοινή πορεία της Ευρώπης. Αυτή είναι η βασική στόχη, να έρθει η Ευρώπη πιο, να γίνει πιο συνεκτική μεταξύ της. Το ΕΦΣΥ δημιουργήθηκε βασικά από τα κράτη-μέλη, είπε ότι έχουμε ανεργία των νέων πάνω από 50% πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Σωστό είναι αυτό. Αλλά όταν ήρθε για το θέμα της χρηματοδότησης Είπαν τα κρατημένα από εμά πεντάρα. Όλα πρέπει να έρθουν από τον κοινό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει απώλεια αλληλεγγύης. Δεν μπορούμε να πούν χρειαζόμαστε τα λεφτά αλλά εμείς δεν θα δώσουμε τίποτα, θα τα δώσετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Οι στόχοι οι οποίοι συνδέονται με το ΕΦΣΥ δεν θα μπορέσουν να επιτευχθούν. Αν δούμε τα σχέδια τα οποία συνδέονται, παραδείγματος χάρη σύνδεση Λιών Τωρίνου με, ένα, με μια σύραγγα. Θα κοστίσει 12 δισεκατομμύρια ενώ το γαλλικό ελεκτικό συνέδριο βλέπει ότι αυτό θα κοστίσει 20 δισεκατομμύρια. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει βέβαια. Και τι θα κόστιζε να ε, αναβαθμίσουμε τις ε, τωρινές γραμμές. Τι θα κόστιζε να κάνουμε καλύτερα τη γραμμή και να αντιμετωπίσουμε τη συναλλαγή. Ενώ τώρα, μα για 20 χρόνια ο, Μετροπό, ο τυφλοπόντικας το μηχάνημα σκάβει της Άλπης, αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει σε κάποια οικονομική ανάπτυξη. Δεν αντιμετωπίζουμε λοιπόν το στόχο της μείωσης ανεργίας με τον τρόπο που γίνεται αυτό. Δεν λέω λέξη βέβαια για κλιματική αλλαγή, γιατί αν αλλάξει, <clears throat> αν υπάρχει αυτή η διαδρομή το τούνελ σε 30 χρόνια, αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου. Επίσης, το τούνελ αυτό περνάει κάτω από την ε, στην Αυστρία ή στις Πανονικές Παιδιάδες. Και πάλι, αν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα, μια ε, γραμμή με ηλεκτρικό τρένο, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης από το τούνελ κάτω από την Αυστρία. Εμείς έχουμε λοιπόν φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουμε κανένα έλεγχο για τα σχέδια αυτά τα οποία είναι κατάλληλα για το ΕΦΣΙ ή όχι εμείς είχαμε αποφασίσει να υποστηρίξουμε ορισμένα προγράμματα παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούσαμε όλοι με όλους αυτά αλλά υπήρχε τουλάχιστον κάποια κοινή συνένεση. Αυτό ήταν σημαντικό. Αλλά μετά δίνουμε τα λεπτά στο εύση και τελείωσε. Δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει τι γίνεται. Μπορεί τώρα το εύση να χρηματοδοτήσει <coughs> ποινικού σταθμού στη Μεγάλη Βρετανία που ο ειδικό τομέα δεν θέλει να το κάνει, αλλά το κράτος είπε δεν υπάρχει πρόβλημα, εγώ για 30 χρόνια θα εγγυηθώ μια τιμή για την ε, ηλεκτρική κιλοβατόρα που είναι τρεις φορές παρά από την αγορά για το πυρηνικό αυτό σταθμό. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με εξοικονόμηση, καμιά σχέση με την ενεργειακή απεξάρτηση, τίποτα απολύτω από όλα αυτά, ούτε βοηθάει την κλιματική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά θα γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και εγώ Βρίσκω τελείως άδικο όχι μόνο να χαναπληρώνω το κοινοβούλιο για όλα, αλλά επιπλέον και αυτό το συζητήσαμε από το συνολικό προϋπολογισμό που εμείς έχουμε στα χέρια μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να ε, προσθέσουμε κάπου χρήματα, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά όταν πρόκειται για μία μείωση για την ε, γεωργία ή κάποιο άλλο τομέα, λένε όχι, αποκλείεται αυτό, δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Λοιπόν, υπάρχει μια απόλυτη έλλειψη αλληλεγγύης. Σε καταστάσεις κρίσης πρέπει να έχουμε μια αλληλεγγύη και τα χρήματα να πάνε εκεί που είναι απαραίτητη η επένδυση και θα βοηθήσει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όχι να λέμε ότι τα δικά μας δικά μας γιατί είναι σημαντικά και για τις μεταφορές δεν θέλουμε να δώσουμε απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν θα ήταν για μένα αλληλεγγύη να θέτουμε κοινού κανόνε, αλλά όχι αυτό το οποίο κάνουμε που διαλέγουμε επιλεκτικά. Εδώ μα βολεύει να πάρουμε λεφτά, εκεί μα βολεύει να πάρουμε λεφτά και έτσι σιγά σιγά απογυμνώνονται οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήμουν ο τελευταίο λοιπόν ομιλητή, πρωτού σα ξαναδώ στο λόγο κύριε Γκάιερ. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ αμέσω σε αυτό που είπες. Δυστυχώς, δεν μπορούμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να πηγαίνουμε από την κατηγορία 1α, ξέρω εγώ, που έχει λεφτά, σε κάποια άλλη. π.χ. ένα Β είναι τα περιφερειακά ταμεία, τρία είναι η πολιτική γεωργία, η άλλη είναι η εξωτερική πολιτική. Δεν άλλα μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά από εδώ να τα πάμε εκεί. Δεν γίνεται. Αυτό είχε κάποτε μια λογική αιτία. Δηλαδή υπήρχε μια εποχή στην οποία ένας γεωργός πληρωνόταν ε, από την ΕΟΚ τότε και είχε εγγυημένη τιμή για το προϊόν του. Και τελικά παρήγαγε όσο περισσότερο μπορούσε και θυμόμαστε τα βουνά από βούτυρο κτλ και χαιρότανε γιατί είχε εγγυημένη τιμή. Για να γλιτώσουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό μπήκαν αυτές οι κατηγορίες και η μεταφορά μεταξύ κατηγοριών πλέον δεν είναι δυνατή για να διατηρηθεί ένα maximum στις γεωργικές δαπάνες. Τώρα ο καιρός αυτός έχει παρέλθει, είναι τελείως διαφορετική η γεωργική πολιτική, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, κάνουμε, δίνουμε μεσεωνικούς αγώνες με το Συμβούλιο όσον αφορά την δυνατότητα απόφαση, απόφασης του Κοινοβουλίου. Βεβαίω ε, μπορεί ο καθένας να πει ότι η κυβέρνησή του, καμία κυβέρνηση σας διαβεβαιώ, δεν θέλει να υποχωρήσει σε οτιδήποτε. Οπότε δεν γίνεται αυτό το οποίο λες να πάρουμε δηλαδή 1% από το, τον κάθε τίτλο και να τα βάλουμε στο Connecting Europe Facility. για να αντισταθμίσουμε το μειονέκτημα του ΕΦΣΗ. Πρέπει να παραμείνουμε εντός της ε, κατηγορίας 1α και εκεί να αναζητήσουμε κονδύλια. Πολιτικά μπορούμε να ζητήσουμε εμείς κάτι άλλο, αλλά Αυτό μετά είναι μια απέτηση που απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Και θα απαιτεί ένα τελείω διαφορετικό κανονισμό για τον προπολογισμό. Να επανέλθω λοιπόν στο μέσο Connecting Europe Facility. Όσο πιο ξεκάθαρη και αποτελεσματική η χρήση των μέσων του Connecting Europe Facility, τόσο καλύτερα τα δικά μας τα επιχειρήματα. Για να προστατεύσουμε τα λεφτά που έχουμε σε αυτό. για να αποδείξουμε ακριβώς τη σημασία που έχει το ΣΕΦ με βάση τα έργα που χρηματοδοτεί, με βάση την οικονομική σημασία που έχουν μετά αυτά τα έργα για τις περιφέρειες και τους διάφορους κλάδους. Για να μπορούμε να έχουμε ορθά επιχειρήματα. Στη διαπραγμάτευση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Για να ε, είναι όσο δυνατόν μικρότερες οι απώλειες και να προστατεύσουμε το Connecting Europe Facility. Και είμαι απολύτως σίγουρος πως η μεγαλύτερη πλειοψηφία εδώ πέρα θα ήθελε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει πλήρως του ΣΕΦ. Οπότε αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου. Αλλά μετά πάμε σε μια διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Και εκεί πέρα θα δούμε το εάν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το Connecting Europe Facility στην έκταση που έχει σήμερα. Να πω όμως κάτι που έχει σχέση με την ε, τρέχουσα συζήτηση. Έχουμε το ΕΦΣΙ, το Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αποδοτικά κερδοφόρα δηλαδή έργα. Έχουμε ένα άλλο μέσο, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Ομόλογα Έργων, που λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, ήταν αν θέλετε το υπόδειγμα για το ΕΦΣΥ, που χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό, δηλαδή το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τουλάχιστον από την Γερμανία αυτό γνωρίζω, χρηματοδοτεί έργα τον αυτοκινητόδρομο Α5 μεταξύ Αμβούργου και Σλέσφιχ Χολστάιν. Και όπως είπαμε έχουμε το Connecting Europe Facility που δίνει επιχορηγήσεις ε, που δεν αναμένουμε ότι θα είναι κερδοφόρες οπωσδήποτε. Αυτό το οποίο με ενοχλεί ειλικρινά είναι το ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιο μέσο χρηματοδοτεί πιο συγκοινωνιακό έργο. Και ε, αν το ξεκαθάριζε κανείς θα ήμουν δύο λέξεις τώρα ακόμα δύο παρατηρήσεις. Θα ξεκινήσω με τον τουρισμό. Την προηγούμενη θητεία ήμουν μέλος της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειακών Θεμάτων. Και όταν συζητούσαμε το πλαίσιο της τωρινής προγραμματικής περίοδου, είχαμε μια, περίοδο, είχαμε μια συζήτηση για το εάν μπορούμε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τουριστικά έργα με το Περιφερειακό Ταμείο. Και αποφάσισε η Επιτροπή μας, όλες οι ομάδες, ότι Μπορεί να γίνει αυτό και πάντα η Κομισιόν έλεγε όταν ζητούσαμε λεφτά για τον τουρισμό ότι αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Ταμείο. Υπάρχει εδώ πέρα λοιπόν μια διέξοδος και εδώ πέρα απευθύνω έκκληση να επιδείξετε κάποια δημιουργικότητα. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, τα πιλωτικά έργα. Αυτή τη στιγμή, στο πλαίσιο του τραν, υπάρχουν 7 πιλωτικά έργα. Κάποια από αυτά έχουν στόχο, ασχολούνται με το θέμα του τουρισμού. Ποιο είναι το νόημα των πιλωτικών αυτών έργων. Σε κάθε προϋπολογισμό υπάρχουν 40 εκατομμύρια ευρώ, όχι παραπάνω, δηλαδή γελίο ποσό, αλλά δεν επιτρέπεται να δώσουμε παραπάνω, για πιλωτικά έργα τα πιλωτικά έργα ε, χρηματοδοτούνται αν πληρούνται δύο όροι. Πρώτον, πρέπει βεβαίω να είναι αρμοδιότητα τη Ένωση, Δεύτερον, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει αυτό το οποίο γίνεται. Πουθενά αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπάρχει ε, χρηματοδότηση για το ίδιο θέμα. Και τότε λαμβάνει την αξιολόγηση Α ένα έργο από την Κομισιόν. Όταν λέω 40 εκατομμύρια, ε, δεν είναι πολλά τα έργα, δηλαδή και 7 είναι πάρα πολλά. Και... Αν θέλετε ο τουρισμός να χρηματοδοτηθεί περισσότερο από τον προϋπολογισμό, απευθύνω έκκληση να σκεφτείτε τα πιλωτικά έργα στον τομέα του τουρισμού και αν είναι επιτυχή θα υπάρξουν κάποια προπαρασκευαστικά μέτρα και μετά αν είναι επιτυχή και αυτά θα υπάρξει ένα πρόγραμμα. Όσα περισσότερα τέτοια επιτυχημένα έχουμε, τόσα περισσότερα επιχειρήματα έχουμε στον επόμενο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό να έχουμε ξεχωριστό προϋπολογισμό για τον τουρισμό. Σας το λέω ειλικρινά δηλαδή, μέσω της τακτικής ε, δημοσιονομικής διαδικασίας ε, δεν θα γίνει. Γιατί μου φέρνουν συνεχώς το επιχείρημα ότι Αυτά θα χρηματοδοτηθούν από, το, από τα περιφερειακά ταμεία. Πρέπει να βρούμε ένα κομμάτι που δεν χρηματοδοτεί το Περιφερειακό Ταμείο και να το ορίσουμε ως πιλωτικό έργο. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι ώστε μέσω πρόθεσμα να έχουμε κάποιες δυνατότητες ευτυχίες. Τελευταία πρόταση με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για τις οποίες εξακολουθώ να είμαι εισηγητής για το θέμα ασφάλειας των ευρωπαϊκών συγκοινωνιών έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρώ πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία περικοπή σε αυτά. Η συγγήτρια το ανέφερε. Αλλά, ε, παραδείγματος χάρη, ναι, επειδή αυτή τη στιγμή η Frontex ε, δεν είναι πλέον συντονιστής ε, των συνοριοφυλακών, αλλά ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή εν τη γενέση, φαίνεται πως οι υπόλοιπες υπηρεσίες πλην της ε, Frontex ε, δεν θα πάρουν πολλά λεφτά. Οπότε ελπίζω να μην έχουν ε, περικοπές αλλά μην περιμένετε και αυξήσεις. Πρέπει να έχετε πολύ καλά επιχειρήματα για το που θα απαιτηθεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και για την ε, συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή και εν καιρό θα ξαναβρεθούμε. Πρωτού περάσω όμως στο επόμενο σημείο τώρα, θα ήθελα να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία της βραζιλιανής κυβέρνησης, η οποία εκτάκτος είναι παρούσα εδώ στην ε, συνάντησή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης και έχω ζητήσει από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει την κατάσταση προετοιμασίας της σε σχέση με τα διευρωπαϊκά σχέδια TEN-T. Ίσως πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην ε, Κομισιόν, εάν θέλει, να μας παρουσιάσει τις τρέχουσες εργασίες της σε σχέση με τα διευρωπαϊκά σχέδια για τους διάφορους ε, διάβολους του κεντρικού δικτύου. Έχουν παρουσιαστεί από τις συντονιστές τα σχέδια εργασίας. Θα θέλαμε τώρα να ξέρουμε ποιες είναι οι περαιτέρω πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κομισιόν για την ολοκλήρωση του δικτύου των TNT. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Ολιβιέ Ονίδη, τον λόγο για μια σύντομη παρουσίαση. Ξέρουμε τώρα ποιοι είναι οι πραγματικοί φίλοι των TNT, αυτοί που μείναν στην αίθουσα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και για να συνδέσω αυτά τα οποία θα πω με αυτά που είπατε στην προηγούμενη συζήτησή σας και επίσης και την πρωινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό θέλω να εκφράσω και πάλι την ε, ε, συγγνώμη μου, έχουμε καταφέρει να βρούμε την επιστολή που έλεγε ο κύριος Πίπας σήμερα το πρωί, η οποία μας έφτασε υπό μορφή ενός email και τώρα έχουμε προετοιμάσει και την απάντηση και η απάντηση πράγματι επιβεβαιώνει αυτά που σας είπα το πρωί. Ποτέ δεν είπαμε ότι δεν θα υπάρξει χρήματο, ότι δεν θα χρειαστεί συμπληρωματική χρηματοδότηση για το ΣΕΦ, για το Connecting Europe. Αντίθετα με απόγνωση ψάχνουμε συμπληρωματικά κονδύλια. Και φυσικά αυτό θα σας το πει και επισήμως η αρμόδια επίτροπος. Αυτή λοιπόν είναι η στάση μας που είναι σαφέστατη. Τεν τι τώρα. Θα ήθελα καταρχήν να ο φόρο τιμή στον ε, κύριο Χάραλ και τους συναδέλφους του που πολύ δεν είναι σε αυτή την αίθουσα γιατί βέβαια η ανάπτυξη του συνολικού δικτύου ξεπερνά πολύ περισσότερο αυτά που ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι από εμά θα περιμέναν όταν εγκρίθηκε ο αρμόδιος κανονισμός. Ξέρω ότι περιμένετε οι συντονιστές να έρθουν να σας παρουσιάσουν όχι μονάχα την ετήσια ε, επισκόψη του έργου της, αλλά και τις προβλέψεις για το έργο στους ε, διαδρόμους, αυτούς τους εννέα διαδρόμους που έχουν εκδηθεί πλέον επίσημα από τα κράτη-μέλη και αυτό ήταν μια όχι μικρού μεγέθους επιτυχία. Όλες οι χώρες δεχτήκανε την ανάλυση και τις συστάσεις των συντονιστών. Και τώρα το εγχείρημα το οποίο μας απασχολεί στα πλαίσια των ten είναι να προχωρήσουμε από μια στατική εικόνα για το τι χρειαζόμαστε στους διαδρόμους αυτούς σε ό,τι αφορά το έργο υποδομής σε μια δυναμική εικόνα του τι χρειάζεται σε επίπεδο επενδύσεων φυσικά αλλά και της προσθήκης στοιχείων που θα οδηγήσουν σε μια τακτική ενημέρωση της κατάστασης των διαδρόμων και την αντιμετώπιση των εμποδίων που πρέπει να έρθουν τα μέτρα για την εφαρμογή αυτών των διαδρόμων που έχουν φτάσει σε ένα βαθμό ορίμων σχεδίων, ημερομηνίε ε, περάτωσης, τα θέματα διαλειτουργικότητα και τα θέματα των τεχνικών προσκομμάτων, όλα αυτά θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Θα καλύψουμε επίσης και μέτρα για τη βελτίωση της χρήση του δικτύου, μέτρα που πολλέ φορές είναι στον χώρο των ρυθμιστικών ή κανονιστικών αρχών, όπως τα θέματα της καινοτομίας και επίσης και δείκτες απόδοσης για να με καταμετρηθεί όχι μόνο ο βαθμό συμπλήρωση των δικτύων αυτών, αλλά και η χρησιμοποίησή τους Και εδώ ερχόμαστε σε ένα από τα θέματα που αναφέρετε σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρο. Με ποιον τρόπο θα κάνουμε τις ε, επιλογές μεταξύ των αρχικών στοιχείων υποδομή που είχαν προβλεφθεί στην αρχή, ενδεχομένως μεγάλων υποδομών, και της δυνητικής αντιμετώπισης του πραγματικού αποτελέσματος των διαδρόμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε άλλες επιλογές με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, ιδίως στις διαμεθοριακές περιοχές των διαδρόμων. Όλα αυτά θα σας τα παρουσιάσουμε στο πλαίσιο των ημερών TNT στο Ρότερνταμ 21 και 22 Ιουνίου. Θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε και την πρώτη συζήτηση, όχι μονάχα με εκπροσώπους αυτής της Επιτροπής, αλλά και με τους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών και με τους άλλους εμπλεκόμενους. Επιπλέον, θα έχουμε τα πρώτα σχέδια για το σχέδιο εργασίας σε οριζόντιο και θεματικό επίπεδο, το έργο για τους ε, λεγόμενους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, όπου ήταν αρμόδιος κάποιος Brian Simpson που γνωρίζετε πολύ καλά και με τον οποίο συνεργαστήκαμε με μεγάλη χαρά. Και επίσης το σχέδιο για το ERTMS και την διαλειτουργικότητα στα συνδρομικά θέματα. Θα έχουμε δύο πολύ σημαντικά εργαλεία λοιπόν εδώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο την εφαρμογή της πολιτικής μας στους δύο αυτούς τομείς επιπλέον, διότι ο Χέραλ δεν έχει ποτέ αρκετή δουλειά και θέλει πάντα και περισσότερη. Έχει ε, φέρει μαζί τους συντονιστές σε μια νέα περιπέτεια. Έχουμε κάνει ένα απολογισμό των σημαντικών συζητήσεων που κάναμε από την έκθεση Μπότβιχ Χριστόφερσον για τη χρηματοδότηση των υποδομών μεταφορών και πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε δεχομένως να εισαγάγουμε και κάποια άλλα ζητήματα με την πρωτοβουλία των συντονιστών και θέσαμε τα εξή πέντε θέματα. Πολυτροπικότητα, ITS το, ITS το FES σύστημα μεταφορών, νέες τεχνολογίες πώς μπορούν να εφαρμοστούν πιο γρήγορα στην αγορά, η διάσταση των αστικών χώρων που είναι πολύ σημαντικά και ποτέ δεν το τονίσουμε αρκετά και εν τέλει η επέκταση των ε, TNT ε, και του πλαισίου τους και σε άλλες χώρες και όχι μόνο τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και σε άλλες. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν στο Ρότερνταμ και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα επανέλθουμε και στην Επιτροπή σας γιατί πολλές από αυτές τις συστάσεις θα θέλαμε να τύχουν συνέχεια είτε με τις εκθέσεις πρωτοβουλία που έχετε προετοιμάσει ή που επεξεργάζεστε ή επίσης σε κάποια νομοθετικά μέτρα που θα κληθείτε να εξετάσετε. Προβλέπονται κάποιες κατεξουσιοδότηση πράξεις. Έχετε μία ενώπιον σας αυτή τη στιγμή που είναι η επέκταση των Τέντη και στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό έχει παρουσιαστεί σε εσά πριν από ένα μήνα περίπου. Και επίσης έχετε το Μάιο μία πρόταση που θα έρθει ενώπιον σας που θα είναι η τεχνική προσαρμογή του πλήρους δικτύου. Έχουμε δει τα στατιστικά στοιχεία και όλα αυτά και θα έρθουμε με μια πρόταση τεχνικής προσαρμογής που θα δίνει τα τελευταία benchmarks για το πλήρες δίκτυο. Τέλος, για τις ημέρες των TNT, ελπίζουμε στο βαθμό του δυνατού να έχουμε στον δυνατόν περισσότερους από την Επιτροπή σας. Θα είναι μια ειδική συνάντηση θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για τα θέματα χρηματοδότησης, γιατί όπως ξέρετε μπαίνουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών και θα είναι και η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια πρώτη αξιολόγηση για όλα αυτά τα οποία έχουμε ενώπιόν μας για τις μεταφορές μέσα στα πλαίσια του ΕΦΣΥ, του προγράμματος επενδύσεων και θα έχουμε και μια ειδική μέρα για να επιτρέψουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι η προαγωγή των σχεδίων αυτών να έρθουν σε επαφή με ιδιωτικούς επενδυτές αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα συζητηθούν τα σχέδια εργασία, τα θεματικά ζητήματα και επίσης θα είναι και η πρώτη ευκαιρία για το σύνολο της οικογένειας των διευρωπαϊκών δικτύων, όχι μόνο οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι υπουργοί των γειτονικών χωρών, ιδίως των Δυτικών Βαλκανίων ή των χωρών της Ανατολικής ε, ε γειτονίας ή της νότιας γειτονίας με την νότια Μεσόγειο και επίσης με την Τουρκία, όλοι αυτοί θα μπορέσουν να συζητήσουν για μας για την περαιτέρω επέκταση των τεντή στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Γειτονίας. Εν τέλει, μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τη σημασία που επέχει η σημερινή συζήτηση. Ξέρω και βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση ότι έχει γίνει αυτή η συζήτηση πριν κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ε, δικιάς σας επιτροπής και χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που έχετε φέρει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και μας έχετε δυνατότητα να κάνουμε αυτή την ειλικρινή ανταλλαγή από Thank you very much as well. Now, Wim ευχαριστώ. Ο Φάντενκαμπ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ο κύριος Πονηδί λοιπόν και η ομάδα του πραγματικά αξίζουν ευχαριστίες για αυτές τις ε, πληροφορίες. Νομίζω πως η Κομισιόν εργάζεται σκληρά, αλλά για το θέμα των διαδρόμων των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ακόμη πιο σκληρά. Και αναμένω τις μέρες διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, που φέτος θα είναι στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία αν δεν το ξέρετε. Ένα από τα ωραιότερα κράτη-μέλη, οπότε χρήσιμο θα είναι αυτό και θα περάσουμε ωραία. Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις. Παρατηρώ εδώ ότι Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ε, χρηματοδότησης για υποτμήματα των διαδρόμων αυτών που αυξάνονται. Έχουμε το ΣΕΦ, το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Συνοχής, Εθνική Χρηματοδότηση. Ε, ε, έχω δικιό, έτσι είναι. Ή δεν υπάρχει αυξανόμενη ευελιξία ως προς τη χρηματοδότηση. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά την Κίνα τι κάνει η Κίνα στις ε, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Είναι μόνο καλά λόγια αυτά ή είναι αυτές οι επενδύσεις ε, στους διαδρόμους κάτι το οποίο ενδιαφέρει την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Ζήνα Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ονιδή για τις εξηγήσει Όλα ωραία ακούγονται. Έχω μία ερώτηση έχω εγώ. Πολλά είπαμε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, νέες τεχνολογίες κτλ. Όλα αυτά ωραία. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως κοινοβούλιο που θεωρούμε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το μέσο συνδέοντα στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά. Τι μπορούμε να κάνουμε για, τα, να τα στηρίξουμε. Δεν ξέρω, ίσως να μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τα στηρίξουμε. Αλλά είμαστε από διάφορες χώρες, έχουμε επαφές με διάφορες κυβερνήσεις. Μπορούμε να πούμε πού είναι τα προβλήματα. Καλό θα ήταν να ξέρουμε. Αν κάποιος έχει στυλώσει τα πόδια κάπου μπορούμε να βοηθήσουμε. αν μου είναι εναντίον κάποιου ευρωπαϊκού έργου και καλό είναι να το ξέρουμε έτσι διμερώς όπως τόσο διπλωματικά λέτε, εν πάση μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ Κάρη Μαντελή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία, παρατήρηση. Τα έγγραφα είναι πολύ πυκνά. Και μας τα στάσκει η Επιτροπή πολύ καθυστερημένα. Αν γίνεται την επόμενη φορά να μας τα πιο νωρίς. Είμαστε εδώ πρόσωπα της Επιτροπής, ε, εσείς και εμείς δεν είμαστε και πολλοί, πάντα μας εντυπωσιάζετε κάθε φορά που ανοίγει το στόμα σας. Να υπενθυμίσω ότι όλοι στην Κομισιόν είναι υπέρ των επενδυτικών έργων, σχεδίων για τις υποδομές. Αλλά ό,τι τι μας είπατε. Μας είπατε ότι πρέπει να δούμε τα project ανάλογα με τους δείκτες επιδόσεων. Ίσως να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά εγώ νομίζω ότι αν έχετε υπόψη στη μεταφορά του 21ου αιώνα, οι επιδόσεις είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Εσείς είπατε μία απίστευτη φράση. Πώς θα επιλέξουμε μεταξύ μεγάλων project και άλλων project. Δεν υπάρχουν άλλα project. Μιλήσατε για την ε, αστική κινητικότητα προτεραιότητα. Ο 21ος αιώνας δεν θα πρέπει να κατασκευάσει τεράστια project, τεράστια έργα ας πούμε, που είναι καταστροφικά για το περιβάλλον, για τους, ε, τις πρώτες κτλ. Όχι κύριέ μου, όλα πρέπει να γίνουν σε τοπικό επίπεδο ο 21 ο αιωνα θα είναι ο αιώνα των μικρών έργων, των έργων γειτονία. Και εδώ δεν κάνουμε πολεμική, ιδεολογική πολεμική ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρηματοδότησε τη γραμμή, ας πούμε, το Τωρίνο. Άλλες γραμμές που χρηματοδότησε η Ευρώπη ήταν καταστροφικές. Παραδείγματος χάρη γραμμή Περπινιό Φιγκέρας, που άρχισε να λειτουργεί το 2009. Ήτανε παλιά πολύ φθηνή, όπου όπου ας πούμε προβλεπόταν ότι θα μετακινούνταν εκεί ε, και πολλοί επιβάτες και πολλά ε, εμπορεύματα ας πούμε. Και όμως δεν την προτιμήσατε, προτιμήσατε το λιό ε, το Ρήνο. Γιατί. Εάν αυτή η Επιτροπή Juncker ε, μια και είπε ο κ. Γιούνκερ ότι είναι η Επιτροπή τη ε, τελευταία ευκαιρία. Εάν δεν τα καταφέρει να συμφιλιώσει του Ευρωπαίου πολίτε με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, καήκαμε. Και στις μεταφορέ, αυτό που μα ενδιαφέρει κυρίω είναι οι αστικέ μεταφορέ. Τι, τι περιμένουμε για να πούμε η βιώσιμη κινητικότητα είναι χρήσιμες επενδύσεις, ε, δημιουργία θέσης ε, έργα καλά για το περιβάλλον, αλλά καλά και για το κλίμα. Ξέρετε ότι, ε, ξέρω ότι θα μου πείτε πως ε, έχω μονομανία με τη γραμμή Λιό-Τωρίνο. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά τα λεφτά τα οποία εξοδεύτηκαν εκεί, ε, τα οποία ήταν αρχικά είχαμε πει 8 εκατομμύρια, τελικά ήταν 12 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει άλλα έργα. Και μάλιστα να εξασφαλίσουν συγκεκριμένες, απτές ανάγκες των πολιτών. Ευχαριστώ, Γιάννης Φρίτς. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από την Βόρεια Σουηδία και έχουμε στενή συνεργασία με τη Φιλανδία στα συγκοινωνιακά για όλες αυτές τις βόρειες περιοχές και μετά υπάρχει και ο άλλος διάδρομος εκεί ο Βαλτικός και θυμάμαι πως κάπου είχα δει μια έκθεση για τη χρηματοδότηση ειδικά των μεγάλων έργων και έλεγε εκεί πέρα ξεκάθαρα ότι όλο αυτό το σύστημα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών πρέπει εξ αρχής να είναι προσανατολισμένο προς το μέλλον. Βεβαίως, ναι, πρέπει να ληφθούν και εθνικές αποφάσεις ε, για να υπάρξει αυτή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εάν αυτές ε, οι αρχές, ε, αυτή η αρχή που ανέφερα εξακολουθεί να υφίσταται. Σας ευχαριστώ. Μαλτέζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Αντέλη έχει μονομανία με τη γραμμή το Ρήνο Λιόν. Και εγώ και εκείνη και ίσως και πρόεδρος Κράμερ. Γιατί. Και διαρωτώ με γιατί και οι υπόλοιποι δεν έχετε αυτή τη μονομανία. Δεν φοβάστε, ε, δεν έχετε ερωτηματικά γύρω από τα μεγάλα ευρωπαϊκά project. Πριν η πράσινη συνάδελφος ε, έλεγε ότι η γραμμή Περπινιό Φιγκέρας κήρυξε πτώχευση, αλλά ήταν μια συνδρομική γραμμή αρχικά που είχε, κόστιζε το ένα έκτο από ό,τι κόστιζε η, η άλλη Λιόν το ε, Ρήνο ε, και όμως και πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία σε επιβάτες και φορτίο. Ε, ξοδεύουμε απίστευτα λεφτά στην Ευρώπη για να φτιάξουμε ένα τερατώδες έργο για, 20 χρόνια και τελικά ε, ξοδεύουμε απίστευτα λεφτά φτιάχνουμε μια γραμμή που είναι πάρα πολύ σύντομη, φτάνουμε στην πόλη που θέλουμε, ε, σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα, αλλά εκεί πέρα κολλάμε στην ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση τη πόλη και χάνουμε απίστευτε ώρε εκεί. Τι νόημα έχει. Στην πράξη, αυτά τα μεγάλα έργα διαψεύδουν όλε τι προτεραιότητέ μα. Όλα όσα λέμε για την επίπτωση στο περιβάλλον, για τη βιωσιμότητα σε οικονομικού όρου, για τη χρησιμότητα των έργων και κινδυνεύουμε να μην μπορούμε να δικαιολογήσουμε τις δράσεις μας ε, στο κοινό. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Είχα μια άλλη παράλληλη συνεδρίαση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το κόστος των μεγάλων έργων υποδομής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι εμείς δεν θέλουμε έργα υποδομών τα οποία κοστίζουν στο Δημόσιο Ταμείο απίστευτα χρήματα και τελικά δεν έχουν καμία αιτιολογία. Δηλαδή δεν εξυπηρετούν τις μεταφορές. Είχαμε πτωχεύσεις ας πούμε που μίλησαν, για τις οποίες μίλησαν ε, οι συνάδελφοι για έργα υποδομών τα οποία δεν εξυπηρέτησαν τους επιβάτες. Αυτά τα έργα δεν δημιουργούν ζήτηση. Συχνά γίνονται αυτά τα έργα, ε, δημιουργείται ένας κύκλος χρήματος ε, γύρω από αυτά, χωρίς καμία διαφάνεια. Εμείς ζητάμε πληροφορίες ε, οικονομικές για αυτά τα έργα για, τις, για τους διαγωνισμούς και τα λοιπά και κανένας δεν μας δίνει αυτές τις πληροφορίες. Η Κομισιόν δεν μας δίνει τα στοιχεία. Όχι μόνο κάποιοι ευρωβουλευτές, αλλά όλο το Κοινοβούλιο στην έκθεση που εγκρίθηκε στην περασμένη σύνοδο στο Στρασβούργο υπερψήφισε την δράση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων μία θέση που λέει ότι θα πρέπει ε, το project το Ρήνο Λιό να διέπεται από απόλυτη διαφάνεια και όχι μόνο αυτό και όλα τα υπόλοιπα έργα υποδομών με ανεξάρτητες αξιολογήσεις για αυτά τα έργα, που συχνά δεν αφορούν το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά μόνο το συμφέρον κάποιων εταιριών και μερικέ φορέ και των εγκληματικών οργανώσεων. Θέλουμε, επομένω, να χυθεί άπλετο φω σε αυτό το έργο. λιον το Και μια και έχουμε εδώ του εκπροσώπου τη Κομισιόν και μια και το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ζήτησε αυτές τις πληροφορίε, ζήτησε αυτή τη διαφάνεια για το έργο Λιόν ε, Θέλω η Κομισιόν τώρα να μου απαντήσει Εάν πρόκειται να δημοσιοποιήσει σε όλους, όπως ακριβώς ζητούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα στοιχεία για το έργο αυτό. Παρακαλώ, θέλουμε να μας δοθούν τα έγγραφα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντέλη. Ο κύριος Ντέλη. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κύριο Ονίδη για την παρουσίασή του και εγώ προσβλέπω επίσης τις ημέρες των TNT στο Ρότερνταμ γιατί ο δικός μου συντονιστής είναι Ολλανδός από το ΕΛΚ και θέλουμε να τον υποστηρίξουμε. Χαιρετίζω λοιπόν τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που μπορούμε να δούμε τα πρώτα λειτουργικά αποτελέσματα της λεγόμενης διαδικασίας του Βερολίνου για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων όπως θυμόσαστε τον προηγούμενο Αύγουστο έγινε μία διάσκεψη στην κορυφή στην Βιέννη και υπήρξαν εκεί συμφωνίες μεταξύ των πρωθυπουργών των χωρών αυτών για τις διαδρομές των διευρωπαϊκών δικτύων και με την επέκταση των δικτύων σε αυτή την περιοχή νομίζω ότι δίνουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για όλη την περιοχή αυτή και την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Να σας αναφέρω όμως και μερικές προτάσεις που θα μπορούσατε να τις λάβετε υπόψη Όπως γνωρίζετε ίσως, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, όπως είναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης των σχεδίων αυτών, για να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα σημεία συμφόρησης και να υπάρξει το θετικό αποτέλεσμα των διαδρόμων στο σύνολο του δικτύου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξανασκεφτούμε για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που δεν ευνοούν τις χώρες αυτές, αλλά αυτό δεν ευνοεί γενικά ούτε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρούνται αυτά τα σημεία συμφόρησης στα Δυτικά Βαλκάνια όταν τα επόμενα δύο-τρία χρόνια σίγουρα δεν θα προχωρήσει πολύ διαδικασία ένταξη των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ε, διεύρυνση της εντολής των συντονιστών των TNT για αυτή την περιοχή και νομίζω ότι με την έγκριση των σχεδίων των TNT θα μπορέσει να ξεπεραστεί αυτό το τυπικό εμπόδιο σε ό,τι αφορά την ε, επέκταση του, της εντολής των συντονιστών ένα τελευταίο στοιχείο πρόσθετο στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας είναι η σχεδιαζόμενη έκθεση για την προσβασιμότητα των υποδομών μεταφορών στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτή η έκθεση έχει προχωρήσει ήδη πάρα πολύ κοντά στο τέλος και στην έκθεση αυτή που έχουμε να σκιωδήσει ήδη από το ΕΛΚ θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Κομισιόν να προχωρήσει στα θέματα της ε, συνδεσιμότητα στην κεντροανατολική Ευρώπη και όπως είπε και ο κύριος Ονίδης θα βοηθήσει και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και χώρες της Ανατολικής Γειτονίας όπως η Ουκρανία να έχουν καλύτερη συνδέση με την Ευρώπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και ο πρόεδρος, ο κύριος Ρίκε. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ονίδη για την ε, πιστή του συμβολή στο έργο της Επιτροπής. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η εξέταση και η οργάνωση των ε, τεντή. Αυτά τα σχέδια σε λειτουργικό επίπεδο κατευθύνονται από μια λειτουργική υπηρεσία αναφορέα της Κομισιόν που έχει ε, ασχοληθεί με αυτό το έργο και που έχει εξουσδιωτωθεί να ξεκινήσει τη λειτουργική χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων και να τα παρακολουθήσει. Τώρα, ποια είναι η σχέση αυτού του φορέα με, το, με την σύνδεση μεταξύ του ΕΦΣΙ, του σχεδίου Juncker και του της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Υπάρχει μια μόνο απευθυντική θηρίδα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εξασφαλίζει ότι αυτοί που καταθέτουν σχέδια να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη μέσα από τις αναλυτικές δομές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για να γίνει η σύνδεση αυτού του λειτουργικού φορέα που έχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των σχεδίων αυτών για τα, μεταξύ αυτής της υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που και αυτή παίζει σημαντικό χαρακτήρα για τις δράσεις ε, συγχρηματοδότησης. Πού λοιπόν υπάρχει η συνεκτικότητα μεταξύ όλων αυτών. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την λειτουργία αυτής της ε, θηρίδας πώς εξασφαλίζεται η συνέχεια δράσης για αυτές τις ενέργειες χρηματοδότηση. Μια, ε, μια δεύτερη παρατήρηση. Εγώ ανησύχησα όταν άκουσα αυτά που είπατε από το κύριο Ανίδη. Αν κάποιος ο οποίος είναι εξίσου ε, εμπειρογνώμων για τα θέματα του προϋπολογισμού της Κομισιόν και μας λέει ότι δεν καταλαβαίνει την διαφορά μεταξύ του ΣΕΦ, του ΕΦΣΙ και των ε, ομολόγων έργου, μα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και αν δεν το καταλαβαίνει αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να εφαρμόσει μια βασική αρχή που είναι η προσεντικότητα και επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημά μου τη σύνδεση μεταξύ αυτών που καταλαβαίνουν καλά στην Κομισιόν Λειτουργικού Φορέας για τα, για τα σχέδια αυτά, αν θα έχουν δημόσιο χαρακτήρα ή σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα νομίζω ότι κατανοούν πολύ καλά την ε, προσθετικότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, ε, συνάφεια μεταξύ των ενεργειών σε επίπεδο προϋπολογισμού και σε επίπεδο λειτουργικό και αυτών που επιθυμούμε εμείς να, να δούμε να γίνεται πραγματικότητα στον τομέα των μεταφορών. Και ένα τρίτο σημείο, αν θέλετε να υπάρξει μια τιτλοποίηση σε επίπεδο ομολόγων έργου και σε επίπεδο εύση των ενεργειών αυτών που γίνεται. Αυτά οι τίτλοι λοιπόν ή τα ομόλογα τα οποία μπορούν να εκδοθούν. Αν υπάρξει λοιπόν τιτλοποίηση για, για, ε, για ενέργειες οι οποίες έχουν μονάχα μία μικρή ε, συμμετοχή του δημοσίου τομέα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί δεν έχει έρθει το θέμα αυτό των, ε, του RTT στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μπιλμπάουδε Μπαραντίκα. Ζητώ συγγνώμη, γιατί και εγώ έρχομαι από μια άλλη συνεδρίαση και δεν μπορώ να είμαι να κλωνοποιηθώ και να είμαι και σε δύο συνεδριάσεις. Τέλος πάντων, Κάποιε από και από τις αμφιβολίες ε, που είχα ε, διατυπώθηκαν ήδη ε, σε σχέση με την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Θα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της, της Κομισιόν, το 2013 κάναμε μία αναθεώρηση των ε, των ε, έργων ε, προτεραιότητας που θα γίνουν μέχρι το 2024. Και όμως το 2016 δεν έχουμε ολοκληρώσει κανένα από τα έργα αυτά προτεραιότητας. σε κάθε κράτος μέλος φυσικά είναι διαφορετική κατάσταση, το ακούσαμε. Θα ήθελα όμως να διατυπώσω δύο ερωτήσεις. Από τη μία, μετά από την αναθεώρηση που έγινε το 2013, με ένα χρηματοδοτικό ε, μέσο, με όλα αυτά τα μέσα που έχουμε και που σχολιάθηκαν, ε, θεωρείται ότι τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής από τα κράτη-μέλη ε, ανταποκρίνονται στα κριτήρια τα αναθεωρημένα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο το 2013 στην αναθεώρησή του. Δεύτερον, ξέρουμε ε, παντού και στην Ισπανία ακόμα και κυρίως στη χώρα των Βάσκων. Υπάρχει ένα κομμάτι του Ατλαντικού άξονα, του άξονα του Ατλαντικού, που την επισκεφτήκαμε στην Επιτροπή Μεταφορών, που έχει ολοκληρωθεί ή μάλλον ένα τμήμα της μόνο και που υπάρχουν διαδοχικές καθυστερήσεις λόγω του ότι δεν χρηματοδοτεί η Ισπανική κυβέρνηση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν έχει γίνει ένας υπολογισμός για το κόστος που υποτίθεται που μας ε, βαραίνει σε εμά τους Ευρωπαίους, ε, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά στη συνοχή, στο περιβάλλον, στο κλίμα κτλ. Πόσο μας κοστίζει η μη εκτέλεση των έργων από πλευράς των μελών. Γιατί συνέχεια μιλάμε για το ότι μας κοστίζει η εκτέλεση, ας πούμε, ότι πληρώνουμε εκατομμύρια, ας πούμε, για έργα. Αλλά αφού ξοδεύουμε να κάρο λεφτά στην αρχή, α πούμε, τι γίνεται όταν ξαφνικά σταματήσουν, ας πούμε, αυτά τα έργα στη μέση και δεν ολοκληρωθούν. Δεν μα κοστίζει και αυτό. Και πόσο μας κοστίζει, θα κάνουμε υπολογισμό. Danke de Αγκούσα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι και η Πορτογαλία είναι ένα κράτος μέρος το οποίο έχει μεγάλη δυνατότητα και ιδίως η περιοχή της Μαδέρα που βέβαια δεν είναι κομμάτι της υπηρετικής μάζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχει και αυτή μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξη. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίασή της εδώ, για το γεγονός μας παρουσίασε αυτό το σχέδιο για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας είναι ένα πρώτο σχέδιο το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ε, ανάγκες και του περιβάλλοντος και έχει συγκεκριμένες γραμμές δράσης. Σχετικά λοιπόν με αυτό το σχέδιο, εγώ προερχόμενη από μια νησιωτική περιοχή της Μαδέρας, Πιστεύω ότι οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας, όπως λέγονται, μπορούν να βοηθήσουν τις περιφερειακές ε, περιοχές της Ευρώπης και τις νησιωτικές περιοχές και επομένως ζητούμε από την Κομισιό να κάνει ό,τι χρειάζεται, ώστε οι νήσοι και οι υπερπεριφερειακές περιοχές να συμπεριληφθούν σε αυτό το σχέδιο δράσης και θα ήθελα να γνωρίσω τι είδου δράσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν για να βελτίσουν την συνεκτικότητα των νήσων μεταξύ τους και με τους διάφορους διαδρόμους. Επίσης πώς θα γίνει η, ο συντονισμός της δράσης του ΣΕΦ με το ΕΦΣΙ και με τα διαφορετικά ταμεία για τα σχέδια τα οποία θα περιλαμβάνουν αυτές τις νησιωτικές ε, και άλλες περιοχές. Αυτά είναι τα ερώτημα τα που θέλω να ζητήσω από την Κομισιόν και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας έχει δώσει στην Επιτροπή μας και που θα είναι πολύ χρήσιμες για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Πάλι έβαλα τον εαυτό μου στον κατάλογο των ομιλητών. Σήμερα το πρωί σας είπα ήδη ότι υποστηρίζω ιδιαίτερα τα τμήματα, τα διαμεθοριακά των τέντι να τύχουν προτεραιότητας και επομένω δεν μπορώ παρά να επενέσω το έργο και τις προτάσεις της Κομισιόν. Πρέπει όμως να κάνω και μερικές επικρίσεις. Έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Υπάρχουν κάποια μικρά προγράμματα και σχέδια τα οποία δεν θα υλοποιηθούν. Πόσο θα κοστίσει αυτό. Το 2014 έκλεισε το χάσμα μεταξύ τα χάσματα μεταξύ, στις συνδύσεις μεταξύ της ε, Γερμανίας και της Τσεχίας. Για λίγες εκατοντάδες μέτρων, χρήσιμο, 650 μέτρα, χρήσιμο, χρειάστηκαν να υπάρξουν 50 χρόνια για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν τα είχαμε κλείσει λοιπόν αυτό πριν από 20 χρόνια και τώρα τα τρένα που κυκλοφορούν είναι γεμάτα, πόσο θα είχε βελτιώσει την κατάσταση. Και η σύνδεση μεταξύ Βερολίνου και Βρότσλαβ και μετά Κρακοβίας, αν είχε ε, εξηλεκτριστεί αυτή η γραμμή. Θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσει ε, δύο ώρες με μονάχα 50 εκατομμύρια όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια για να κάνουμε το ίδιο σε σχέση με τη σύνδεση Τωρίνο-Λιών. Τι θα είχαμε κερδίσει λοιπόν και πόσο γρήγορα θα τα είχαμε αποσβέσει αυτά ενώ για την σύνδεση Λιών-Τωρίνο μάλλον δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα αποσβέσουμε. Αλλά λέω για το Λιόν Τωρίνο, γιατί ήμουνα στο τελευταίο ταξίδι της ε, αντιπροσωπείας μας στη Λαπωνία και στο ε, Ελσίνκι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον δήμαρχο του ε, Ελσίνκι. Λέει ότι και εμείς θέλουμε να ανήκουμε καλύτερα στην Ευρώπη και να έχουμε ένα τούνελ υποθαλάσσιο από το Ελσίνκι στην Ταλίν. Αυτό ήταν το όνειρό του και είπε αυτό, ναι, πρέπει να έχουμε και τα μέσα συνοχής τη Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότηση 40%. Και σκέφτομαι τώρα για το Τωρίνο. Αντί να κάνουμε αυτό το τούνελ, θα μπορούσαμε να κάνουμε το τούνελ Ταλίν Ταλήν-Ελσίνκη. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας θέσω αυτό το ερώτημα, δεν πρόλαβα να το κάνω το πρωί. Αν υπάρχουν κάποιε ε, κάποιοι υπολογισμοί αν εξηγιανθούν και αναβαθμιστούν οι τωρινέ συνδέσεις πόσο θα κοστίσει και πόσο θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Και αυτό έγινε για τη γραμμή τωρινού Λιών, όταν στην αρχή λέγαμε ότι θα ήταν 12 δισεκατομμύρια το κόστος, αλλά το Γαλλικό Ελεκτικό Συνέδριο και η Γαλλία το υποστηρίζει αυτό, μας είπε ότι είναι 26 δισεκατομμύρια το κόστος. Μήπως υπάρχουν τώρα νέοι υπολογισμοί πόσο θα κόστιζε αυτό σε σχέση με την εξυγίανση απλώ του υπάρχοντος δικτύου και την δημιουργία θέσεων απασχόληση που θα προέκυπτε. Θα ήθελα λοιπόν πολύ καλά να ξέρω με ποιο τρόπο έγινε ο υπολογισμό αυτό για τα 12 δισεκατομμύρια και μετά αν έγινε νέο υπολογισμό ή όχι, αν μπορείτε τουλάχιστον να μας κάνετε μια σύγκριση για τα παλιά αυτά στοιχεία που είχατε. Και μου είπαν επίσης στο τελευταίο σημείο ότι θα περάσει από το ε, υψίπεδο των, από, τις από την πανονική πεδιάδα μάλλον μια, ένας νέος διάδρομος. Και προτιμούν να περιμένουν να περάσει αυτή η σύνδεση από, τη δική τους από δικό τους μέρος α, και όχι να παρακάμψει την περιοχή αυτή. Αυτό θα έχει μεγάλη επίπτωση στον διάδρομο μέσω των πανονικών του παρονικού υψηπέδου και αν γίνει κάτι τέτοιο αντί για ένα μία σύραγγα αυτό θα βελτιώσει πολύ περισσότερο την κατάσταση γιατί το τούνελ θα έχει πάντα έλλειμμα. Σε, γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να περνάνε πάντα τα μεγάλα σχέδια όσο πολυδάπανα και να είναι ενώ τα μικρότερα σχέδια τα αφήνουμε στο περιθώριο. Σα ευχαριστώ. Έχετε θέσει, λοιπόν, έχουμε θέσει λοιπόν πολλά ερωτήματα και περιμένουμε με αδειμονία την απάντησή σα κύριε Ονίδη. Thank you. Thank you, That was Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι πολλές οι ερωτήσεις. Να προσπαθήσω να τι απαντήσω με την σειρά. Είχαμε τι ερωτήσει του κυρίου Φαντεκάμπ. Νομίζω τα σχέδια εργασίας δεν θα δώσουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Αλλά τουλάχιστον ε, θα δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια στο τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ποια πηγή. Η κυρία Μάισνερ ρώτησε ειλικρινά τι μπορείτε να κάνετε ως βουλευτές να συνεχίσετε να στηρίζετε την ε, διαδικασία ε, έτσι ώστε να υπάρχουν ακριβώς οι πτυχές της ε, χρηματοδότησης που χρειαζόμαστε αλλά βεβαίως ο γεγονός είναι πως ακόμα έχουμε κάποιες αποφάσεις ασυνάρτητες δηλαδή εθνικές επιλογές που δεν συμφωνούν με τις προτεραιότητες που είναι πιο λογικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξακολουθούν να μην είναι βέλτιστες οι επιλογές όσον αφορά τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται. Δεν λέω ότι μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό ή να πειθαρχήσουν όλοι, αλλά τουλάχιστον με την δεύτερη αυτή γενιά έργων θα έχουμε όλα τα στοιχεία επιτάπτως για να υπάρξει αυτή η κριτική ανάλυση και μια συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω πως και στην δική σας την ε, περιφέρεια και με τις διάφορες επαφές που έχετε στο πολιτικό επίπεδο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με βέλτιστο τρόπο το υλικό που υπάρχει σε αυτά τα σχέδια εργασίας για να γίνει πιο λογική επιλογή. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Όσον αφορά την Κίνα, νομίζω ότι ορίζουμε οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης. Η Κίνα έχει μεγάλη ρευστότητα, αλλά η Κίνα κατά κύριο λόγο ενδιαφέρεται σε κάποια έργα όπου η χρηματοδότηση δίνεται όταν ε, πληρώνονται κάποιοι όροι. Δηλαδή να χρησιμοποιεί κανείς κινέζικο εξοπλισμό, εργολάβους, να κάνει παραχώρηση για 50 χρόνια κτλ. Αυτά δεν γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ακολουθήσει τους ίδιους κανόνες με τους άλλους επενδυτές και έχουμε τώρα αυτόν τον διάλογο στη λεγόμενη πλατφόρμα σύνδεσιμότητας ε, με την Κίνα και ελπίζω εκεί να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους Κινέζους ε, εταίρους μας ε, ποιοι είναι οι κανόνες και είμαστε πολύ ειλικρινείς και βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Ένα συμβολικό που υπεγράφει πρόσφατα ε, σιδηρόδρομος Βελιγραδίου Βουδαπέστης που έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι όροι ε, που είχαμε διαπραγματευτεί φαίνεται πως δεν ε, συμμορφώνται πλήρως με τους όρους περί δημοσίων προμηθειών. Τα συζητάμε λοιπόν με τις Ουγγρικές και Σερβικές αρχές και με τους Κινέζους καθώς βλέπουμε πως ασκείται πίεση ειδικά στις πιο ευπαθείς χώρες που ετοιμάζονται να ενταχθούν στην Ένωση αλλά δεν έχουν πει ακόμα και χρειάζονται επενδύσεις υποδομών. Οπότε... Βλέπουμε ακριβώς τι προτεραιότητες υπάρχουν μπροστά μας. Και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο το Λιόν Τωρίνο και πολλά άλλα έργα, αλλά εντός αυτών των ε, έργων τα στοιχεία αυτά υπάρχουν, τα γεγονότα επίσης είναι διαθέσιμα και είμαι στην διάθεσή σας για να σας δώσω όλες τις πληροφορίες που ίσως θέλετε για να αναλύσετε το χ, το ψ έργο για το Λιόν Τωρίνο. Μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε κριτική θέλετε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν έχει διαφάνεια. Κανένα άλλο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ελεγχθεί τόσο πολύ και δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο τόσων πολλών συζητήσεων. Αυτό το δέχομαι. Αντιλαμβάνομαι πως βλέπετε με, κριτικό, με κριτική, επικριτική σκοπιά το θέμα αυτό, γιατί δεν το θεωρείτε ίσως το σημαντικότερο έργο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα μέτρα που οδήγησαν τον νομοθέτη και το Κοινοβούλιο να επιλέξουν αυτό το συμβολικό έργο για τις οριζόντιες πτυχές ε, νομίζω πως ε, το τονίσατε και ελπίζω να μπορέσουμε τελικά να περιλάβουμε στην περιγραφή των υποδομών και στοιχεία του τι μπορούν να αποτελέσει υποδομή η θα είναι πιο έξυπνη, πιο πράσινη κτλ. Και εδώ πέρα κοιτάμε όλα τα θέματα που εξετάζουμε στα θεματικά μας έγγραφα για να χρησιμοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τους πένιχρούς μας πόρους. Ναι, τώρα το ερώτημα του κυρίου Νίλσεν για την, τα, χρηματοδότηση. Ναι, πράγματι, ακριβώς αυτό γίνεται για να ξεκινήσουν τα έργα σε πολύ δύσκολες φάσεις Οπότε τα έργα τα οποία στηρίζουμε είναι πράγματι ε, έργα τα οποία δίνουμε σημαντικά ποσά στην αρχική φάση. Δεν τα εγκαταλείπουμε μετά. Αλλά, όπως σας είπα, η περισσότερη χρηματοδότηση δίνεται στην αρχή. Όσον αφορά την επέκταση του πλαισίου των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Χαίρομαι ιδιαίτερα όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά το ότι ανήκει και σε άλλε γειτονικέ χώρες. Νομίζω πως ε, αυτή η δικτύωση είναι αυτό ακριβώ το οποίο προσπαθούμε να αναλύσουμε και στο έγγραφο που έχουμε για την εξωτερική διάσταση. Ελπίζουμε να έχουμε κάποιο χρήσιμο υλικό για τους συναδέλφου μας ε, που είναι αρμόδιοι για την ε, οικονομική στήριξη στις χώρες αυτές για να γίνουμε δικά τους μέσα. Αλλά βλέπουμε ότι όλες αυτές οι χώρες είναι αρκετά πειθαρχημένες για να Ε, επιδείξουν κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και βεβαίως να υπάρχουν και κάποιες ρυθμιστικές αλλαγές ε, για να υπάρξει μετά στη ατζέντα των ήπιων μέτρων που λέμε για να έρθουν σιγά σιγά κοντά στο κοινοτικό κεκτημένο. Το, η νέα τώρα δεν εμπλέκεται αμέσως ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά σαφώς είναι ένα κέντρο αριστείας όσον αφορά τη γνώση των διαφόρων έργων. Γνωρίζετε τη συζήτηση που έχουμε τακτικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οφείλουμε να σεβαστούμε την εξαρτησία της τράπεζας και της Διαχειριστικής Επιτροπής της ΕΦΣΕ, νομίζω πως στο επίπεδο εργασίας έχουμε συνεχείς άμεσες επαφές με την Τράπεζα Επενδύσεων και η ΙΝΕΑ ακριβώς ε, τροφοδοτεί το κομμάτι εκείνο το οποίο είναι αρμόδιο για τις μεταφορές. Γιατί όπως ξέρετε δεν λειτουργεί ακόμα στο 100% και δεν έχουμε μια ομάδα ειδικών για τις μεταφορές. Οπότε χρησιμοποιούμε όλους τους πόρους, ε, την Κομισιόν, την ΙΝΕΑ ε και τους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Τώρα, για την αιρεσιμότητα υπάρχει και στο χρηματοδοτικό τομέα και μπορούμε να πούμε ναι ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν χρειαζόμαστε επιπρόσθετους πόρους. Είναι απλοποιημένη αυτή η προσέγγιση και έχουμε στις μεταφορές ειδικά επιδείξει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ε, χρηματοδοτικά μέσα υπό τον όρο, ή υπό τον όρο για περίπλοκες περιπτώσεις ότι θα υπάρχει επιπρόσθετη στήριξη υπομορφή επιχορηγήσεων. Οπότε παρακαλώ να είστε στο πλευρό μας Στι δύσκολες συζητήσεις που θα γίνουν για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, αλλιώς ε, γρήγορα θα καταλήξουμε σε μία ε, ακριβώ ε, προσέγγιση για όλους. Για την τιτλοποίηση κάποιων έργων δεν έχουμε ακόμα φτάσει εκεί γιατί δεν υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χαρτοφυλάκιο παρόμοιων έργων. Μια πραγματική τιτλοποίηση θα μπορούσε να υπάρξει όταν θα έχουμε κάποια θεματικά χαρτοφυλάκια, πηχιαστικά έργα, λιμενικά έργα που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κάποια τέτοια μέσα. Και τέλος, είναι πάντα δύσκολο να διαλέξουμε ημερομηνία για τις μέρες διευρωπαϊκών δικτύων. Έχουμε, όπως είπαμε, ακριβώς ε, αυτή την ε, σύγκρουση που υπάρχει. Ελπίζω λοιπόν να έρθετε μαζικά και οπωσδήποτε ελπίζω να έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις πριν ξεκινήσει η Ολομέλεια. Σημειώνω επίσης τις παρατηρήσεις της κυρίας Μπιλμπάου και του Προέδρου. Νομίζω πως είναι ένας πολύ καλός τρόπος αυτός ε, είναι για να επανατοποθετηθούμε όσον αφορά το τι χρειάζεται και ποιες είναι οι προτεραιότητες. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε με βάση τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή να δούμε έργα πολύ περισσότερο με τον τρόπο που περιγράψατε, δηλαδή να αναλύσουμε το κόστος, τις συνέπειες της μη χρηματοδότησης αυτών των έργων. Γιατί έχετε δίκιο εδώ, ούτε ένα έργο πρώτης προτεραιότητας του παλιού καλού καιρού δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Κοιτώντας λοιπόν τις διαφορετικές επιλογές και προτεραιότητες, νομίζω ότι μια τέτοια ανάλυση θα μας βοηθήσει να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε κάποιες από τις ε, αλλαγές προτεραιοτήτων που θα κάνουμε. Δεν λέω ότι θα έχουμε το τωρινό παράρτημα του κανονισμού του συνδέοντας στην Ευρώπη ως έχει. Εγώ είμαι ο πρώτος που θέλω να αλλάζει αυτό με τρόπο δυναμικό, ε, με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και ίσως ε, να δούμε ε, πού θα πάει χρηματοδότηση, πού θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Κυρία Μοντέρα, η αυτοκινητόδρομη της θάλασσας, χαίρομαι που έχουμε η επιτέλους κάποιες εξελίξεις για αυτό το σημαντικό και περίπλοκο θέμα. Κατ' ουσίαν έχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν οι πρώτες μέρες, δηλαδή προσπαθήσαμε να μετακινήσουμε στο δυνατόν περισσότεροι συγκοινωνία από τους δρόμους στην θάλασσα και αυτό είναι ο βασικός μας στόχος υπό την ηγεσία του Μπραν Σίμψον και η δεύτερη πτυχή είναι η σχέση με τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Αυτή ήταν νομίζω η υπόσχεση τότε. Είπαμε πως ε, δεν ε, υπάρχει, δεν υπάρχουν αυτό, δεν είναι πολύ τονισμένες αυτές οι πτυχές, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα για να συνδέσουμε τα νησιά και άλλες απομονωμένες περιφέρειες. Και αυτό θα τονιστεί στο σχέδιο εργασίας του κ. Σίμψον. Τέλος, συμπερασματικά, Νομίζω πως ε, έτσι είναι αυτή η αντιμετώπιση των ε, διαδρόμων θα μας βοηθήσει να έχουμε όλες αυτές τις επιλογές και εσείς βεβαίως θα είστε μέρος αυτής της συζήτησης και θα χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα που υπάρχουν, ε, τα έγγραφα των διαφόρων θεμάτων, τα σχέδια εργασίας, πάρα πολύ καλές αναλύσεις με όλα τα νούμερα, με ανάλυση, χαρακτηριστικά των ε, μέσων μεταφοράς για να μας βοηθήσετε να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε... Ευχαριστώ, αλλά δεν απαντήσατε σε κάποια ερωτήματα. Σας ρώτησα αν υπήρξε μια νέα ανάλυση μετά από την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας που είπε ότι θα κοστίσει 26 δισεκατομμύρια και όχι 12 και αν δικαιολογείται αυτή η αύξηση 14 δισεκατομμύρια. Και τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει ο νέος διάδρομος από την Πρατισλάβα ως τη Μεσόγειο, υπήρξε μια νέα ανάλυση για το τούρελ που θα τη συνοδεύει, τη στιγμή που υπάρχει ήδη το η διαδρομή αυτή η οποία είναι ήδη πολύ χρήσιμη για τις εμπορευματικές μεταφορές αν έχει νόημα να υπάρξει αυτή η νέα σύνδεση με σύραγγα. Υπάρχει λοιπόν μια νέα αξιολόγηση και έχετε τα στοιχεία για αυτήν ή όχι. Ευχαριστώ. Που επαναφέρεται στην τάξη που με αναγκάζει να απαντήσω στις ερωτήσεις που προσπαθώ να αποφύγω. Για το Λιό Τωρίνο. Έγινε μια ανάλυση για τα όσα είπε το γαλλικό ελεγκτικό συνέδριο, επιβεβαίωσε το αρχικό κόστος με την προσθήκη βέβαια του πληθωρισμού. Έχουμε φτάσει τώρα στα, σε ένα συνολικό κόστος 12 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή το νούμερο που έδωσε το γαλλικό ελεκτικό συνέδριο δεν είναι σωστό. Ε, για το δεύτερο ερώτημα με ξεπερνάει. Ε, δυστυχώς θα πρέπει να σε απαντήσω γραπτός. Ε, δεν εντάξει είμαι γενναιόδωρος, θα σας δώσω αυτή τη δυνατότητα. Ο κύριος Ρικέ. Να απαντήσω εγώ στο ερώτημα. Διαφορά, για τη διαφορά αυτή που είχαμε για το Λιόν Τωρινό. Τα 9 δισεκατομμύρια Συν την ε, υποτίμηση κάνουν 12. Το σχέδιο χρηματοδότηση βασιζόταν στο γεγονός ότι υπήρχαν πολλά τούνελ. Πρέπει να φτάσουμε στα τούνελ. Τα 14 αρχικά δισεκατομμύρια χρειάζονται για να φτάσουμε στο πρώτο τούνελ και από εκεί πέρα προστίθονται και άλλα ποσά για το υπόλοιπο έργο. Ο κύριος Φάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνει δυνατότητα να δευτερολογήσω. Δεν μου αρέσει το στυλάκι της Κομισιόν. Όταν σας ζητάμε πληροφορίες, η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών που ανήκω, πήρε μια απόφαση να δοθούν αυτές οι πληροφορίες σε σχέση με αυτό το έργο το Ρήνο Λιών. Έχουμε στείλει και ένα έτοιμα από τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι δηλαδή τη ομάδα μου, αλλά από όλο το Κοινοβούλιο, για να έχουμε αυτέ τι πληροφορίε, ενώ η Γενική Διεύθυνση μου δεν μα απαντάει. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει διαφάνεια, να χυθεί το φω, να μα δώσετε πληροφορίε. Δεν μπορείτε να μα λέτε ότι υπάρχει ήδη διαφάνεια. Δεν υπάρχει. Θέλουμε το συντομότερο δυνατόν αυτέ τι πληροφορίε και δεν ξέρω αν εσεί μπορείτε να μου τι δώσετε. Θέλω τέλο πάντων μια και το αίτημα αυτό δεν είναι δικό μου, δεν είναι από κάποιε πολιτικέ ομάδε, αλλά από όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μα δώσετε, εν πάση περιπτώσει, αυτέ τι πληροφορίε ή αλλιώ να μα δώσετε το γιατί, και αυτό να είναι δημόσιο, δεν μπορείτε να μα παράσχετε αυτέ τι πληροφορίε που σα ζητάμε επιτακτικά. Έδωσα τη δυνατότητα σε τρει ε, ομιλητέ να θέσουν τα ερωτήματα και φυσικά και εσεί έχετε τώρα δυνατότητα να απαντήσετε για το τελευταίο σημείο, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα είμαστε πάντα μαζί σας και θα σας δίνουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχουμε. Πάντα θέλουμε να σας δίνουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια αυτά. Ό,τι μας ζητάτε θα το δίνουμε. Εκτός, εκτός, εκτός φυσικά, αν η προαγωγή των σχεδίων μας ζητούν να μην αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες. Αλλά αυτό ισχύει μονάχα για μερικά από τα έγγραφα που είναι το τμήμα της επίσημης πρότασης και τεκμηρίωσης που βρίσκεται στα αρχεία μας. Όλο το υπόλοιπο όμως, η αναλύση, η λογιστική έλεγχη, όλα αυτά είναι δικά σας. Θα έχετε πρόσβαση σε αυτά και με μεγάλη ευτυχία θα έρθουμε να σας συναντήσουμε ακόμα και διμερώς για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την παρουσίασή σας, για τις απαντήσεις που δώσατε στα ερωτήματά μας. Ήταν μια ζωντανή και πολύ καλή συζήτηση και φυσικά θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα θέματα αυτά. Τα, το επόμενο θέμα δεν βλέπω τίποτα στα διάφορα. 5-7 Απριλίου στις 9 η ώρα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας και ούτως έχει τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση και χαίρομαι που μπορούμε να τα ξαναπούμε στις 7 Απριλίου. Ευχαριστώ πολύ και καλή μέρα σε όλους.